Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους ε, που παρήθανται, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν μέσω ε, σύνδεσης. Θα ήθελα στην έναρξη της συζήτησης να εκφράσω κάποιες σκέψεις ε, για τα θύματα του κορονοϊού, ε, προς τις οικογένειές τους, προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και θα ήθελα σε όλους τους ασθενείς ε, να ευχηθώ ταχύτατη ανάρρωση. Αυτή τη στιγμή το υγειονομικό προσωπικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά του συγκεκριμένου ιού και αξίζουν όλη την υποστήριξή μας, το θαυμασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας για ε, τη δουλειά που κάνουν και για την γενεοδορία με την οποία τους διακρίνει ε, για ε, ε, την αντιμετώπιση αυτών των ε, καταστάσεων που πολύ συχνά είναι δραματικές. Και βεβαίως ε, και για όλους τους εθελοντές και το προσωπικό που υποστηρίζουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το είπα και το επαναλαμβάνω, η ανθρωπιά των πολιτών μας είναι ο μεγαλύτερός μας πλούτος. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους ε, τους εργαζομένους που ε, κρατούν ε, σε λειτουργία την κοινωνία μας. Τους γεωργούς, τους υπαλλήλους, όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται στις τηλεπικοινωνίες, τους ανθρώπους ασφαλείας, οι ένοπλες δυνάμεις, οι ταμείες των σούπερ μάρκετ η τεχνική των γραμμών που μας επιτρέπουν να συνδεόμαστε, να μπορούμε να τηλεφωνούμε, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ε, ενεργοί στο τομέα της αρμοδιότητάς τους και με πειθαρχία και αίσθηση ευθύνη δεν ε, εγκατέλειψαν. Για όλους αυτούς φυσικά ε, μόνο ένα ευχαριστώ μπορούμε να πούμε και φυσικά δεν θα πρέπει να λησμονούμε και όλους εκείνους τους πολίτες ε, που με πολύ απλές χειρονομίες ε, δείχνουν ε, ένα διαφορετικό τόνο. Σέβονται τα προληπτικά μέτρα. αγοράζουν για έναν ηλικιωμένο γείτονα τα ψώνια του, ίσως διατροφικά προϊόντα. τηλεφωνούν σε απομονωμένους φίλους και φροντίζουν τους πιο ευάλωτους από εμά. Μικρές χειρονομίες ε, συγκεκριμένης αλληλεγγύη. Όπως άλλωστε προσπάθησε να ε, επιδείξει αλληλεγγύη και το δικό μας το κοινοβούλιο ε, διαθέτει τις κουζίνες του για την Παρασκευή χιλίων γευμάτων την ημέρα και πραγματικά αυτά δίνονται στους εθελοντές και τα κτίρια μας στις Βρυξέλλες θα φιλοξενήσουν 100 ευπαθείς γυναίκες αλλά και στο Στρασβούργο και στο Λουξεμβούργο διαθέσαμε στις αρχές τα κτίρια του Κοινοβουλίου για δραστηριότητες που αφορούν αυτή την επίγουσα ανάγκη. Είναι οι πόλεις που μας φιλοξενούν και σε αυτές οφείλουμε ε, ιδιαίτερη αναγνώριση και θα ήθελα μαζί σας να χαιρετήσω και τους πολίτες των Βερξελών, του Στρασβούρου και του Λουξεμβούργου και να πω ότι πολύ σύντομα ε, θα είναι πολύ ευχάριστο να ξανασυναντηθούμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για την Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριότητες του ε, Κοινοβουλίου δυστυχώς ε, χτυπήθηκαν από την επίγουσα ανάγκη και ομολογώ ότι βρέθηκαν να αναλάβω δύσκολες πρωτοβουλίες αλλά πάντα με υποστήριξαν και με ενθάρρυναν όλες οι πολιτικές ομάδες. Καμία ομάδα εξαιρουμένης και ε, άκουσα και συμβουλές πάρα πολλών ευρωβουλευτών. Βεβαίως η λειτουργία του Κοινοβουλίου δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την έκτακτη υποστήριξη και εξαιρετική υποστήριξη του προσωπικού και της διοίκησης μας ε, οι οποίοι με θάρρος και αίσθηση καθήκοντος ε, ήταν παρόντες ε, και φυσικά όλοι οι, γενικές όλοι οι γενικοί διευθυντές ήταν εκεί. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει την ευγνωμοσύνη μας στους εργαζομένους οι οποίοι ίσως είναι και αυτοί που είναι πιο κρυμμένοι οι άντρες και οι γυναίκες της Υπηρεσία καθαρισμού και της υπηρεσία ασφάλειας ε, αλλά και όλοι εκείνοι που στο προσωπικό των γενικών διευθύνσεών μας ε, μας επέτρεψε να ε, μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις μας. Οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμα και να παραμείνει ανοιχτό και να λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με όλα τα όργανα, αποδεικνύει ότι εμείς τα θεσμικά όργανα είμαστε σε θέση να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας. Και θέλουμε να ε, πριτανεύσουν οι αξίες μας ακόμα και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η δημοκρατία δεν σταματά. Πρόκειται για χαλεπούς καιρούς και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Και να σκεφτούμε και βαθιά την κοινωνία η οποία μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο ε, θα ζει διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεσμεύεται ήδη πλήρως για να ικανοποιήσει τις απαιτήσει των πολιτών και των κρατών μελών προς το συμφέρον τους, προς το κοινό συμφέρον μας και στη διάρκεια αυτής της κρίσης ε, αλλά και στη συνέχεια ε, θα είμαστε ακόμα εκεί στο πλευρό τους γιατί εμείς θέλουμε να βγούμε πιο ισχυροί από αυτή την κρίση, πιο εύρωστοι και να είμαστε περισσότερο σε θέση να αντιμετωπίσουμε αύριο τις προκλήσεις που θα μας παρουσιάσει ο παγκόσμιος ε, ο κόσμος μας. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να διαθέσουμε και υγειονομικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα και φάρμακα ε, βασικά, να υποστηρίξουμε την έρευνα και να βοηθήσουμε και να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, να υποστηρίξουμε οικογένειες, ε, τους φτωχότερους και φυσικά να παράσχουμε βοήθεια στους γεωργούς, τους αλληλείς, τους επιχειρηματίες, τους εργαζομένους Μόνο από κοινού μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα για το καλό των πολιτών μας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συντονίσουμε τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων περιορισμού και να βγούμε από αυτή την κρίση. Συμφωνούμε λοιπόν με την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστώ και την Πρόεδρο για την παρουσία της εδώ, διότι θέλουμε να βγούμε από την έκτακτη ανάγκη με τακτικό και συντονισμένο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε και ε, παλινδρομήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι και καταστροφικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις δημοκρατίες μας και να ακούσουμε τους πολίτες μας. Τους ε, ερετούς εκπροσώπους που έχουμε δει σήμερα θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό ψήφισμα για τη συντονισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της ε, καθώς φυσικά και κάποια άλλα εκτακτά μέτρα. Η δέσμευσή μας είναι να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις για τα καλύτερα μέτρα τα οποία θα πρέπει να αναλυφθούν και να ε, αναθέσουμε φυσικά και τα κατάλληλα κονδύλια τα οποία θα πρέπει να διαθέσουμε στα κράτη-μέλη ώστε να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, διότι οι πολίτες μας, οι Ευρωπαίοι πολίτες, ε, περιμένουν από εμά γρήγορες απαντήσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είμαστε η φωνή των πολιτών και πρέπει να είμαστε περήφανοι ε, αυτή τη στιγμή διότι συμβάλλουμε με πειθαρχία για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι και να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε τους λαούς μας για ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Με την έκτακτη σύνοδο συνεχίζουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεκόπη στις 26 Μαρτίου. Εγκρίνουμε τα πρακτικά τα οποία έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Κάποιες ανακοινώσεις, αναθεώρηση του ε, ημερολογίου του 2020 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στην τελευταία συνεδρίαση της Διασκέψης των Πρόεδρων 5η 2 Απριλίου αποφάσισα μαζί με τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων να συγκαλέσω τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση, η οποία συνεχίζεται και αύριο 16 και 17 Απριλίου, ωστόσο, ώστε να ψηφίσουμε τα νέα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση του COVID-19 και να συζητήσουμε την επικαιροποίηση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώ θα καταπολεμηθεί η πανδημία και οι συνέπειε τη. Το προσωρινό ημερολόγιο που αναθεωρήθηκε για το 2020 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μα ανακοίνωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης. Ε, το τελικό σχέδιο ημερησίας διάταξης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Θα ήθελα ωστόσο να σας ενημερώσω ότι έλαβα 10 ε, διαδικαστικά αιτήματα δυνάμει του άρθρου 163 του ιστορικού κανονισμού για να προσθεθούν τα ακόλουθα νομοθετικά έγγραφα και δημοσιονομικά έγγραφα που σχετίζονται με την επιδημία COVID-19 και τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν κατά την ολομέλεια αυτή, την τρέχουσα ολομέλεια. Τροποποιητικός κανονισμός για το πολιτισμό σε νομικό πλαίσιο 2014-2020 Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 1 κάθετος 2020. Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 2 κάθετος 2020 κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020, κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020 2056, κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες δαπάνες για το 2020, ειδικά μέτρα για την παροχή ευελιξίας εξαίρεση για τη χρήση των διευθυντικών ταμείων και των επενδυτικών ταμείων η εισαγωγή ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19, ειδικά μέτρα για το μετριασμό των συνεπειών της επιδημίας ε, COVID-19 στον τομέα της αλίας και των διαδοκαλλιεργειών, ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και κατά συνέπεια μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να ε, θέσω ε, στην Ολομέλεια τις ακόλουθες προτάσεις τροποποίησης του οριστικού σχέδιο ημερήσια διάταξη, δηλώσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή ε, για την ε, ε, καταπολέμηση τη πανδημία. Η συζήτηση θα λάβει χώρα από τι 9, από τώρα δηλαδή, μέχρι τι 12. Το πρόγραμμα των γύρων ψηφοφοριών για την 5η 16 Απριλίου και την Παρασκευή 17 Απριλίου έχει ω εξή. πρώτο γύρο ψηφοφοριών θα ανοίξει από τι 9.30 μέχρι τι 10.30 με τι ψηφοφορίε για τι παραπάνω διαδικασίε ε, επίγουσες διαδικασίες και για το πρώτο μπλοκ τροπολογιών για την πρόταση κοινή ε, κοινοψηφίσματος για την συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πανδημίας. Η Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου ψηφοφοριών προβλέπεται για τη 1.30. Δεύτερο γύρο ψηφοφοριών θα ανοίξει στη 1.30 έω τι 2.30 με μια ψηφοφορία για τον κανονισμό που τροποποιεί το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και για το δεύτερο μπλοκ τροπολογιών για την πρόταση ψηφίσματος, κοινή πρόταση ψηφίσματο για την συντονισμένη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη πανδημία COVID-19 και των συνεπειών τη. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου προβλέπεται βλέπετε για τις 5 το απόγευμα. Ο τρίτο γύρος ψηφοφοριών θα ανοίξει στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 6 με ψηφοφορίες για το τρίτο μπλοκ τροπολογιών για την πρόταση ε, κοινού ψηφίσματος για τη συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και τι συνέπειε. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου γύρου προβλέπεται για τις 8 και μισή. Ο τέταρτο γύρος ψηφοφοριών θα ανοίξει στις 8 και μισή μέχρι τις 9 και μισή με ψηφοφορίες για το τέταρτο μπλοκ τροπολογιών για την πρόταση πρόταση κοινού ψηφίσματο για την συντονισμένη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη πανδημία COVID-19. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα λάβει χώρα στι 10 και 50, 11 παρα 10 το η νύχτα και θα κλείσει η Ολομέλεια στις 11. Αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσει η Σύνοδος στις 9 με τον πρώτο γύρο ψηφοφορίων από τις 9 μέχρι τις 10 και οι ψηφοφορίες για τροπολογίες που σχετίζονται με τα εξή κείμενα σχέδιο διορθωτικού πολυπολογισμού 1 καθώς 2020 και σχέδιο διορθωτικού πολυπολογισμού 2 2020. Άλλη ψηφοφορία, δύο έγγραφα για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020. Τρίτη ψηφοφορία για το έγγραφο για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτα περιστατικά. Τέταρτο, τρία έγγραφα συναπόφασης για το Corona Package 2 και ιατροτεχνολογικά μηχανήματα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προβλέπεται για τις 12.30. Ο δεύτερος γύρος ψηφοφοριών θα ανοίξει στις 12.30 μέχρι τη 1.30 με τελικές ψηφοφορίες για σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 1 και σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 2. Δύο έγγραφα για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020. Έγγραφο για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτα περιστατικά. Τρία έγγραφα συναπόφασης για το Corona Package 2, ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και κοινό ψήφισμα για τη συντονισμένη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη πανδημία και των συνεπειών τη. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει προβλεφθεί για τι 4 το απόγευμα. Τρίτο γύρο ψηφοφοριών για τροπολογίε και τελική ψηφοφορία για μια επακόλουθη πρόταση ψηφίσματο για τον COVID-19 θα μπορούσε ενδεχομένω να λάβει χώρα μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στι 7.30 αύριο το βράδυ. Τέταρτος γύρο ψηφοφοριών για τροπολογίε ή τελική ψηφοφορία για μία επακολουθή πρόταση ψηφίσματο για την πανδημία και τι συνέπειές τη, θα μπορούσε ενδεχομένω να λάβει χώρα από τι 7.30 μέχρι τι 8.30 αύριο το βράδυ με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 10.30 αύριο το βράδυ. Θα κλείσει η Σύνοδος Ολομέλειας στις 11 αύριο το βράδυ. Υπάρχουν ενστάσεις, όχι, οπότε η τροποποίηση εγκρίνεται. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε 9.30 σε λίγο δηλαδή θα ανοίξω τον πρώτο γύρο ψηφοφοριών. Θα είναι ανοιχτό ο γύρο ψηφοφορίων από τι 9.30 μέχρι τι 10.30. Όλε οι ψηφοφορίε τη σημερινή μέρα θα γίνουν με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορούν να επαληθεύσουν την ψηφοφορία του και τα αποτελέσματα οι ευρωβουλευτέ στο έγγραφο, το οποίο θα δημοσιευτεί σήμερα στην ιστοσελίδα τη Ολομέλεια. Και πάμε τώρα στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού, Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών και δίνω το λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Σαρλ Μισελ. Έχετε το λόγο. Έχετε παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι Ευρωβουλευτές. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφραστώ σήμερα σε αυτήν την ε, εξαιρετικά σημαντική συζήτηση για να μπορέσει να ζει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία να αναπνέει ακόμα και σε αυτές τις εξαιρετικές, εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Και βεβαίως ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προς αυτούς και αυτές που άμεσα ή έμεσα έχουν πληγεί από αυτή την κρίση, από αυτόν τον ιό που χτυπάει την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Και να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς όλους τους πολίτες ιδίω στην Ευρώπη που έχουν κινητοποιηθεί έχουν αποδεχθεί τον περιορισμό τόσο σημαντικών ε, κεφαλαιόδων ελευθεριών που μας αγγίζουν όλους. Σε μια στιγμή σαν και αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία. Η μόνη επιλογή είναι να βοηθήσουμε ένα τον άλλον μεταξύ πολιτών, μεταξύ χωρών, μεταξύ περιοχών του κόσμου. Αυτό είναι που διαπνέει τη δράση μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες για να σας δείξω πώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με τα κράτη-μέλη προσπαθεί να λάβει τις ευθύνε του. Είχαμε τρία Ευρωπαϊκά Συμβούλια μέσω βιντεοδιάσκεψης αφιερωμένα στην κρίση του κορονοϊού για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε καθημερινά το συντονισμό των δράσεων, τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η πρώτη φιλοδοξία μας όταν αντιληφθήκαμε το μέγεθος της κρίσης ήταν να μπορέσουμε να μετριάσουμε τη διάδοση του ιού. Δηλαδή ενθαρρύναμε τη λήψη μέτρων με περιορισμούς στα σύνορα που βεβαίως επηρεάζουν την λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μια κινητοποίηση για να βοηθήσουμε τους ε, ερευνητές μας έτσι ώστε να βρεθούν θεραπείες, να βρεθούν εμβόλια. Προσπαθούμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κινητοποιήσουμε ε, πόρους. Ε, υπάρχει και μία προσπάθεια για να συγκεντρώσουμε πόρους. Ε, έτσι ώστε σε επιστημονικό επίπεδο να βρεθούν λύσεις ε, σε επίπεδο θεραπείων και εμβολίων. Θα ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένος ε, και πολύ ευθύ. Διπλή είναι η εντολή που έδωσε το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να δουλέψουμε πάνω σε έναν οδικό χάρτη που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες συστάσεις, σε κάποιες αρχές βέλτιστων πρακτικών για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών όταν θα περάσουμε στη φάση εξόδου, στη στρατηγική προοδευτική εξόδου από αυτά τα περιοριστικά μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, με διάφορα βέβαια επίπεδα περιορισμού. Το δεύτερο σκέλος είναι να προτείνουμε στους αρχικούς κρατών κυβερνήσεων μια κοινή στρατηγική έτσι ώστε προοδευτικά ε, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα να αναπτύξουμε στρατηγικές οικονομικής ανάκαμψης αλλά και οικονομικής αλλαγής. Θα πρέπει στο μέλλον να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να συνεργόμαστε περισσότερο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ποια είναι κατά την άποψή μου τα τέσσερα κεφάλαια για τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσει μια συζήτηση και να παρθούν κάποιες αποφάσεις από κοινού κάποια βήματα από κοινού. Η πρώτη προτεραιότητα κατ' εμέ για να μπορέσουμε ε, να φέρουμε σε πέρα αυτή τη στρατηγική είναι το θέμα της ενιαίας αγοράς. Πώς μπορούμε να επιδιορθώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, αν θέλετε, την ενιαία αγορά ε, και πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε, να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά ταυτόχρονα. Διότι αυτή είναι η πρώτη μας μεγάλη δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν ε, το Ευρωπαϊκό Green Deal, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα ε, να μην πάψουν να είναι οι πρώτες προτεραιότητες. Είναι ένας πολύ σημαντικός μοχλός για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί τα επόμενα χρόνια. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να χτίσουμε μια πολύ ισχυρή βιομηχανική στρατηγική και ταυτόχρονα να εξετάσουμε ε, να δούμε μάλλον τι θα γίνει με το τεράστιο δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να οικοδομήσουν μια ισχυρή στρατηγική για το μέλλον. Πιστεύω επίσης ότι το θέμα της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να ε, αναπτυχθεί περαιτέρω. Υπάρχουν ε, ήδη προτάσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσε που έχουν συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η ισχύ αυτή τη ευρωπαϊκή αγορά, αυτή η δυνατότητα τη ε, κυκλικής ε, οικονομία και τη ανάπτυξή τη, ε, τη αντιμετώπιση τη κλιματικής αλλαγής, τη ψηφιακής ατζέντα, όλα αυτά θα μας δώσουν και μεγαλύτερη στρατηγική ανεξαρτησία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν ο ευρωπαϊκός, ε, ο διεθνής ρόλος της Ευρώπης πρέπει και, αυτός να ληφθεί υπόψη. Πρέπει ε, όλοι να συμμετάσχουμε για να έχει αυτήν την σημαντική διεθνή διάσταση ο ρόλος της Ένωσης. Επίσης πρέπει να αναπτύξουμε μια πολύ ισχυρή στρατηγική για να επενδύσουμε, να επενδύσουμε μαζικά. Ε, με εθνική, υπάρχει μια εθνική διάσταση, υπάρχει όμως και μια ευρωπαϊκή φιλοδοξία εδώ. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να φτάσουμε σε μια συμφωνία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί μακρόν τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίου μήνες για αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα Ίσως όμως να είναι και μια μοναδική ευκαιρία η επόμενη, τα επόμενα 7 χρόνια πώς θα μπορέσουμε με αυτόν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό να δώσουμε κάποια εργαλεία, κάποιες δυνατότητες ε, για την ανάπτυξη αυτής της ισχυρής στρατηγικής που χρειαζόμαστε για το κοινό μας μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Πριν από μερικές εβδομάδες, ε, πριν την κρίση του κορονοϊού, είχα ζητήσει ε, να αυξηθεί το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να αυξηθούν οι δυνατότητές της μόχλευσης ε, και επικέντρωσης ε, σε συγκεκριμένες επενδύσεις. Και βεβαίως εδώ υπάρχει ένα στοιχείο, μια διάσταση αλληλεγγύης που συνδέεται και με την εσωτερική αγορά, διότι πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όλα τα κράτη-μέλη, όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν να έχουν την ίδια φιλοδοξία να πετύχουν και να έχουν τα μέσα για να το πράξουν αυτό και να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω, και είναι πολύ σημαντικό και αυτό, είναι η εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωπολιτική φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τι αξίε μα, τα συμφέροντά μα, τα οποία αυτή τη στιγμή πλήττονται τι τελευταίε εβδομάδε. Και βεβαίω, σε αυτό το ζήτημα τη εξωτερική δράση, εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στη σχέση μα με την Ήπειρο την Αφρικανική. Με, με άλλου πολλού Ευρωπαίου ηγέτε και Αφρικανού ηγέτε, τι τελευταίε ώρε μπορέσαμε από κοινού να εκφράσουμε κοινέ φιλοδοξίε, βραχυπρόθεσμε αλλά και μεσοπρόθεσμε, να υποστηρίξουμε περισσότερο τα υγειονομικά συστήματα ε, στην Αφρική, να ανοίξει αυτή η συζήτηση του χρέου ε, που πραγματικά επιβαρύνει και δυσκολεύει τη δράση των Αφρικανικών κυβερνήσεων και θα πρέπει πιο μέσω μακροπρόθεσμα να έχουμε και μια επένδυση, ε, μια φιλοδοξία μάλλον έξυπνων επενδύσεων ε, σε μια εταιρική σχέση με τις χώρες αυτές που να σχετίζονται και με το Green Deal, να σχετίζονται και με την ψηφιακή ατζέντα. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι εδώ ε, έχουμε κοινά συμφέροντα. Υπάρχει μια αντικειμενική συμμαχία εδώ την οποία πρέπει να ενεργοποιήσουμε του επόμενου μήνε, τα επόμενα χρόνια. Και το τέταρτο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι αυτή η απέτηση πλέον να τεθεί το θέμα τη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και το θέμα της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας. Πώς θα μπορέσουμε τελικά να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από αυτή την κρίση για να είμαστε πιο ισχυροί αύριο οι διαδικασίες λήψη αποφάσεων να βελτιωθούν, οι διαδικασίες συνεργασίας να βελτιωθούν. Ε, αυτά που ανακοινώθηκαν και που συζητήθηκαν, αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, ενδεχομένως τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, όταν θα έχουμε και τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, αυτό θα, αυτό θα είναι ο πολιτικός χώρος, ο δημοκρατικός χώρος, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά για να μπορέσουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες, από όπου και αν προέρχονται, να συμμετάσχουν σε αυτήν την κοινή φιλοδοξία. Πώ θα μπορέσουμε λοιπόν και από κοινού να τλήσουμε κάποια διδάγματα και τέλο, στα πλαίσια αυτή τη φιλοδοξία ε, να μπορέσουμε ε, να πετύχουμε μια στρατηγική ανάκαμψη, μια στρατηγική αλλαγή, οι αξίε τη ε, ένωση, τη αλληλεγγύη, τη ελευθερία, τη ενότητα πρέπει να είναι σημεία αναφορά. Πρέπει να είναι ένα φάρο που μα δείχνει το δρόμο. Διότι αυτή την κρίση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, αυτή την κατάσταση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε Πρέπει να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με βάση αυτές τις αξίες τις ευρωπαϊκές. Αυτός είναι ο κινητήριος μοχλός για μας. Είναι πολλές λοιπόν οι προκλήσεις. Η ευρωπαϊκή ιστορία μας έχει δείξει ότι όταν αντιμετωπίζουμε τις πιο δύσκολες καταστάσεις, εκείνη τη στιγμή που φαίνονται ανυπέρβλητα τα εμπόδια, εκείνες λοιπόν τις ίδιες στιγμές βρίσκουμε τις, δυνάμεις ε, για να βοηθήσουμε ένα τον άλλον να έρθουμε πιο κοντά, να επιδείξουμε δημιουργικότητα, θα χρειαστούν όλα αυτά. Στην Ευρώπη προφανώ υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, διαφορετικέ ιδέε, διαφορετικέ ευαισθησίε για το τι πρέπει να γίνει μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά εγώ είμαι πεπισμένο ότι με ένα πνεύμα αισιοδοξία, με ένα πνεύμα αποφασιστικότητα και με αυτό την, την βούληση να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό δημοκρατικό πνεύμα, να λειτουργήσουν τα θεσμικά όργανα που είναι αυτά που εγγυώνται αυτή ε, τη δημοκρατία, θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε εμεί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είμαστε σε διαρκή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστούμε για αυτό το σχέδιο ψηφίσματο που ε, πλαισιώνει πολύ ορθά ε, το έργο το οποίο θα πρέπει να διαρριχθεί το επόμενο, το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα 27 κράτη-μέλη ε, θα συμμετάσχουν έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουμε προς αυτή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, άρχεται η ψηφοφορία για τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία και δίνω το λόγο στην πρόεδρο Φοντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, Ευρωβουλευτές, δεν υπάρχουν ε, καλά λόγια για να μιλήσουμε για τον πόνο της Ευρώπης ε, και για το πόσο υποφέρει ο κόσμος. Η σκέψη μας είναι σε όλα τα θύματα, αλλά προσευχόμαστε και όλες, για όλες τις οικογένειες που έχουν πένθος. Ε, υποσχόμαστε να διηγηθούμε τις ιστορίες τους και να ε, θυμηθούμε τη ζωή τους και τις μνήμες τους ε, και να μην ξεχάσουμε κανέναν από αυτούς. Θα θυμόμαστε τη Ζουλή, την νεαρή Γαλλίδα που είχε όλη τη ζωή μπροστά της και το Γιάν, ένα Τσέχο ιστορικό ο οποίος πάντα έδινε μάχη για τις αξίες του. Ή ακόμα και τον Τζίνο, τον Ιταλό γιατρό ο οποίος ε, διέκοψε τη σύνταξή του για να βοηθήσει τη... και να σώσει τις ζωές των άλλων. Θα θυμόμαστε την απίστευτη θυσία της ε, Σουζάν που άφησε τον αναπνευστήρα για τον πιο νέο στο Βέλγιο και την εικόνα του Φράνσις ο οποίος χαιρέτησε τον αδερφό του μέσα από το παράθυρο του νοσοκομείου στην Ιρλανδία. Θα θυμόμαστε την ε, νέα ε, Πολωνή μητέρα η οποία δεν θα δει το παιδί της να μεγαλώνει και το νέο ε, ποδοσφαιριστή της Ισπανίας ο οποίος δεν θα δει τα όνειρά του να πραγματοποιούνται. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Τις μητέρες, τους πατεράδες, τις αδελφές, τους αδελφούς τους νέους, τους αγαπημένους ανθρώπους από το βορρά, από τον νότο, από την Ανατολή, από τη Δύση, τους φίλους τους συναδέλφους, ε, τους γείτονές μας ε, και τους ε, ξένους που βλέπουμε στο πεζοδρόμιο. Ανθρώπους που έχουν πράγματα να μας πούνε και πράγματα να δουν και φυσικά από αυτούς τους ανθρώπους εξαρτάται η αγάπη μας. Ε, κάθε μία από αυτές τις δεκάδες χιλιάδες ιστορίες ε, πραγματικά ε, παίρνει ένα μικρό, μια μικρή θέση στην καρδιά μας. Αλλά φυσικά παιρνει μικρο μια μικρη θεση στην καρδια μας αλλα φυσικα ειναι και η αποφασιστικότητά μας η οποία εντείνεται για να μπορέσει η Ευρώπη να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να ζω, ε, σώσει όλο και περισσότερες ζωές. Αξιότιμα μέλη δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιος μια πανδημία που εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα και σε τέτοια κλίμακα χωρίς την αλήθεια. Χωρίς την αλήθεια για τα πάντα, για τα στοιχεία, για τα επιστημονικά επιστημονικά δεδομένα, για την πρόβλεψη, αλλά φυσικά και τις δικές μας τις πράξεις. Ναι, πράγματι, κανένας δεν ήταν προετοιμασμένο στην πραγματικότητα για κάτι τέτοιο και είναι γεγονό ότι πολλοί δεν ήταν παρόντε εγκαίρω όταν η Ιταλία χρειάστηκε βοήθεια στην αρχή. Και ναι, ε, Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σωστό η Ευρώπη να ε, δώσει μια βαθιά συγνώμη για την Ιταλία. Αλλά το να πούμε απλώς συγνώμη έχει αξία αν αλλάξει και συμπεριφορές. Και η αλήθεια είναι ότι ε, πολύ σύντομα όλοι συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να προστατεύσουμε αλλήλως, πρέπει να προστατευτούμε. Και η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη πλέον έχει γίνει ε, ο παλμός της αλληλεγγύης παγκοσμίω. Η πραγματική Ευρώπη λοιπόν υψώνει το ανάστημό τη. Η Ευρώπη που είναι δίπλα στους υπαλλήλους όταν χρειάζεται περισσότερο. Αυτή όπου υγειονομικό προσωπικό από την Πολωνία και γιατροί από τη Ρουμανία σώζουν ζωές στην Ιταλία, όπου αναπνοηστήρε από τη Γερμανία δίνουν ε, συνέχεια στη ζωή στην Ισπανία. Όταν ε, ε, οι γιατροί από τον Πέργαμο πηγαίνουν στις κλινικές στη Βόνη. Βλέπουμε ιατρικό εξοπλισμό να πηγαίνει από τη Λιθουανία στην Ισπανία και αναπνευστήρες να πηγαίνουν από τη Δανία στην Ιταλία. Πράγματι λοιπόν είδαμε ε, οποιοδήποτε ιατρικό εξοπλισμό να πάει προς πάσα κατεύθυνση στην Ευρώπη για όσους έχουν περισσότερους να τους δώσουν σε αυτούς που χρειάζονται. Και αυτό πραγματικά με κάνει περήφανη που είμαι Ευρωπαία. Βεβαίω υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δακτυλοδεικτούν και να κατηγορούν ακόμα και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα προτιμούσαν να μιλούν απλώ ω λαϊκιστέ ε, και να πούνε τη λαϊκιστική αλήθεια. Σε αυτού πρέπει να πω φτάνει. Σταματήστε και ε, να έχετε το σθένο να πείτε την αλήθεια. Να έχετε το σθένο ε, να σταθείτε στο ύψο των περιστάσεων. Γιατί η ένωσή μα είναι αυτή η οποία θα μα βοηθήσει να τα ξεπεράσουμε και θα είναι μια ισχυρή Ευρώπη ακριβώ όπω θα τη διαμορφώσουμε σήμερα και αν χρειάζεστε έμπνευση, Απλώς δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι λαοί ε, στέκονται μαζί ο ένας με τον άλλον με ε, ταπεινοφροσύνη, με ανθρωπιά και πραγματικά αποτείω φόρο τιμή σε όλους αυτούς τους ε, οδηγούς ε, delivery, τους courier, ε, τους, τα μία στα μαγαζιά, αυτούς οι οποίοι αλλάζουν την παραγωγή τους, τη γραμμή παραγωγής για να κατασκευάσουν εξοπλισμό που χρειαζόμαστε, οι Πορτογάλοι εθελοντές οι οποίοι ράβουν μάσκες για τους γείτονέ τους ή τον 7χρονο Έλληνα πιανίστα ο οποίος συνέθεσε ένα τραγούδι για να δώσει θάρρος στους ανθρώπους. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ και αποτείω φόρο τιμή στου ήρωέ μα, στο ιατρικό προσωπικό, τη νοσοκόμα, ε, του ανθρώπου που φροντίζουν άλλου. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ε, μελανιέ στο πρόσωπό του και τραγικέ εικόνε ε, στην καρδιά και στο μυαλό του. Αυτοί οι άνθρωποι που κρατούν το χέρι των ασθενών με ε, αφοσίωση και αγάπη διότι δεν μπορούν να είναι και οι οικογένειε τους. Είναι αυτοί οι οποίοι σώζουν τις ζωές μας και σώζουν ε, και την τιμή μα. Πρέπει λοιπόν να τους προστατεύσουμε ώστε να μπορέσουν να μας προστατεύσουν όλους. Και τώρα θα επικεντρωθούμε στο δρόμο που θα μας δοηγήσει στο να εξοπλιστούμε επαρκώς ιατρικά στην έρευνα για ένα εμβόλιο. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθούμε για να μπορούμε να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα αγαθά και γι' αυτό έχουμε μια ομάδα από τους καλύτερους εμπειρογνώμονες, άντρες και γυναίκες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ζουν, χρησιμοποιούν τη γνώση τους για να σώζουν ζωές. Θα πρέπει λοιπόν, ε, γι' αυτό ε, καταργούμε το ΦΠΑ από τα ιατρικά μηχανήματα που εισάγουμε από τρίτες χώρες και πρέπει να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση που έχουμε δώσει Κάθε διαθέσιμο ευρώ που έχουμε πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε να φανταστούμε για να σώσουμε ζωές, για να προστατεύσουμε τις ζωές των Ευρωπαίων. Γι' αυτό προτείναμε ό,τι μέσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τον σημερινό προϋπολογισμό να τα βάλουμε σε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης. Μιλάμε για περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάνε κατευθείαν εκεί που είναι απαραίτητα για αναπνευστήρε, για προστατευτικό εξοπλισμό, για περισσότερα τεστ, για ιατρική βοήθεια, για του πιο αδύναμους και για εκείνους που αναμένουν μέσα στους καταβλισμούς προσφύγων. Γι' αυτό προτείνουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικά Ταμεία να τα χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση της κρίσης κορώνα. Να δώσουμε δηλαδή πλήρη ευελιξία μπορούν τα μέσα αυτά να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιφέρειες, εκεί που είναι πιο αναγκαία, ανεξαρτήτως από τις ε, όρους που είχαμε με τη συγχρηματοδότηση και τις δεσμεύσεις. Με αυτό το πακέτο, για το οποίο θα ψηφίσει σήμερα το σημερινό κοινοβούλιο, η Ευρώπη υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων της. Και η ίδια αρχή ισχύει και για την προστασία των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων. Η Ευρώπη έχει ξαναντιμετωπίσει οικονομικές κρίσεις, αλλά ουδέποτε κλείσαμε οικονομικά με αυτόν τον τρόπο. Κανείς δεν πρέπει να κατηγορηθεί. Όλοι θα χρειαστούν υποστήριξη. Χρειαζόμαστε μέτρα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό ώστε η οικονομία μας να μπορέσει να ανακάμψει το συντομότερο δυνατόν. Και εδώ πάλι πρέπει οπωσδήποτε να πούμε την αλήθεια. Είναι σημαντικό. Η Ευρώπη έχει κάνει περισσότερα τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες από ό,τι έκανε τα τέσσερα πρώτα χρόνια της προηγούμενης κρίσης. Οι κανόνε μα έχουν γίνει πιο ευέλικτοι από ποτέ. Τι τελευταίε μέρε έχουμε εγκρίνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις, 1,2 δισεκατομμύρια για τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ελλάδα και ε, εκατομμύρια για Πορτογάλους ε, ε, ψαράδε. Έχουμε παραδείγματα για τη Λετωνία, για την Εστονία, για το Βέλγιο, για τη Σουηδία. Για πρώτη φορά στην ιστορία μα ενεργοποίησαμε την πλήρη ευελιξία και το σύμφωνο σταθερότητας με τα μέτρα που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρασχεθεί ε, δημοσιονομική δύναμη άνευ προηγουμένου και η απόφαση της περασμένης εβδομάδας από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης σημαίνει ακόμα περισσότερα δισεκατομμύρια ευρώ για όλους όσους τα χρειάζονται. Στο πλαίσιο όλων αυτών εγώ παροτρύνω όλα τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν στο μέγιστο όλα αυτά τα σχέδια που προτείνει η Κομισιόν για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους από τον κίνδυνο της ανεργίας. Θα παρέχουμε 100 ε, δισεκατομμύρια ώστε τα κράτη να μπορέσουν να καλύψουν ε, σε περίπτωση που μειώθηκαν οι ώρες εργασίας σας ή αν μείνατε άνεργοι και χρειάζεται βοήθεια. Είναι διπλό το όφελος Πρώτον, θα βοηθήσουμε του ανθρώπου να πληρώσουν του λογαριασμού του, τα ενίκια του, τα φαγητό του και να διατηρηθούν και επιχειρήσει ζωντανέ στην όλη διαδικασία. Και δεύτερον, αποτελεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αυτή καθεαυτή το κράτη-μέλη που θα μπορέσουν θα δημιουργήσουν διασφαλίσεις ούτω ώστε οι άλλοι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν εκείνους, να βοηθήσουν εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο στις χώρες τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης η συλλογική απάντηση της Ευρώπης ανέρχεται σε πάνω από 3 3-3 εκατομμύρια ευρώ. Ουδέποτε έχει υπάρξει τέτοια ανταπόκριση τόσο εντυπωσιακή πουθενά στον κόσμο. Αλλά όπως γνωρίζουμε θα χρειαστούμε περισσότερα, πολλά περισσότερα διότι όλο αυτό θα διαρκέσει πολύ και ο αυριανός κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός από τον χθεσινό. Αξιότιμα μέλη, είμαι πεπισμένη ότι η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει αυτόν τον νέο κόσμο. Εάν συνεργαστεί και ανακαλύψει ξανά το πρωτοπόρο της πνεύμα. Και γι' αυτό θα ήθελα να παραθέσω μια πρόταση που είχε γραφτεί από δύο από τους μεγαλύτερους οραματιστές της Ευρώπης ε, και της Ιταλίας, Ελτήρος Πινέλη και Αρνέστο Ράση. Ένας από τους ε, ιδρυτικούς μας πατέρες που έγραψαν από τα κοιλιά της φυλακής τους ένα απομακρυσμένο νησί στην έξαρση του πολέμου όπου είχε χαθεί κάθε ελπίδα για μια ενωμένη Ευρώπη. Τότε αυτοί μας είπαν τα εξή παρηγορητικά λόγια. Έχει έρθει η στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να απορρίψουμε όλα τα παλιά μας βάρη, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για τον νέο κόσμο, ο οποίος έρχεται, ο οποίος θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που είχαμε φανταστεί ποτέ. Αγαπητοί φίλοι, έχει έρθει η στιγμή ξανά να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας χώριζε, ό,τι μας έκανε να τσακωνόμαστε και να λιλοκατηγορούμαστε, να βγούμε από τις ταμπορωμένες μας θέσεις, να πάμε στον νέο κόσμο, για τον οποίο είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλη μας τη δύναμη, το πνεύμα μας και τη δύναμη του κοινού μας στόχου. Αφετηρία θα πρέπει να είναι η κοινωνία μας, οι κοινωνίες μας, οι οικονομίες μας να γίνουν πιο ανθεκτικές. Για να βρούμε απαντήσει σε αυτό το νέο κόσμο χρειάζεται θάρρος, εμπιστοσύνη, αισιοδοξία και αλληλεγγύη και θα χρειαστούν μαζικές επενδύσεις για να μπορέσει να επανακινηθεί η οικονομία μας. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Marshall για την ανάκαμψη της Ευρώπης το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί αμέσως αυτή τη στιγμή. Μόνο ένα εργαλείο έχουμε, το οποίο εμπιστεύονται όλα τα κράτη-μέλη που ήδη υπάρχει και το οποίο μπορεί να παρέχει γρήγορα αποτελέσματα, είναι διαφανές, και έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν ως εργαλείο συνοχής, σύγκλησης και επενδύσεων. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα αποτελέσει την αυαρχίδα της ανάκαμψής μας. Γι' αυτό το λόγο ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι διαφορετικός από ό,τι είχαμε αρχικά φανταστεί, όπως είπε ακριβώς ο Σπινέλη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη όλου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες επενδύσεις που χρειαζόμαστε για να επανικοδομήσουμε την ενιαία αγορά μετά τον κορώνα. Θα παρέχουμε προκαταβολικές πληρωμές ούτως ώστε να ενδυναμώσουμε αυτές τις επενδύσεις τα πρώτα χρόνια της ανάκαμψης γιατί αυτή η κρίση είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη έχουμε δει. Πλήττει σοβαρά υγιείς επιχειρήσεις διότι έχει κλείσει η δημόσια ζωή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καινοτόμε λύσει ε, στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να ξεκλειδώσουμε μαζικέ ιδιωτικέ και δημόσιε επενδύσει, ώστε να επανεκκινήσουμε τι οικονομίε μα και να μπορέσουμε να ανακάμψουμε προ μια πιο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο υποστηρίζουμε, αλλά να διαμορφώνουμε τι βιομηχανίε μα, τι υπηρεσίε μα για να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Θα πρέπει να επενδύσουμε στις ψηφιακέ τεχνολογίε, στις υποδομέ, στην καινοτομία, όπως ε, τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανεξάρτητοι και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις νέες ευκαιρίες. Επίσης σημαίνει το να διπλασιάσουμε τη στρατηγική μας ε, ανάπτυξη επενδύοντας σε αυτήν καθώς θα επέλθει η παγκόσμια ανάπτυξη, ανάκαμψη, η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν θα επιβραδυνθεί. Θα πρέπει να βρούμε τα σωστά σχέδια για να αντιμετωπίσουμε τα κλιματικά προβλήματα. Μια πιο σύγχρονη, μια πιο κυκλική οικονομία θα μας απελευθερώσει από διάφορες εξαρτήσεις και θα μας κάνει πιο ανθεκτικούς. Αυτό πρέπει να μάθουμε από την κρίση. Το να επενδύουμε σε μεγάλη κλίμακα στην καινοτομία, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις καθαρές μεταφορές, ε, στη ε, βιώσιμο τρόπο ε, διατροφής και στην αποκατάσταση της φύσης θα μας βοηθήσει περισσότερο από ποτέ. Αυτό είναι καλό όχι μόνο για τις οικονομίες μας και το περιβάλλον μας. Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε οποιασδήποτε εξαρτήσεις θα έχουμε πιο μικρές αλυσίδες προμηθειών και πιο διαφορετικές. Και κάτι άλλο πρέπει να μην ξεχνάμε. Η κρίση μπορεί να είναι συμμετρική, αλλά η ανάκαμψη όχι, διότι ο ιός δεν είναι το μόνο που έχει πλήξει το οικονομικό σοκ σε ορισμένες περιοχές ε, θα ανακάμψει και σε άλλες θα είναι πιο δύσκολο. Έτσι λοιπόν η σύγκληση και η συνοχή θα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Η ενιαία αγορά και η πολιτική συνοχή είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Χρειαζόμαστε και τις δύο για να έχουμε ευημερία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμα μέλη. Αυτή η Ευρώπη πιστεύω μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από αυτή την κρίση. Αυτή που κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τι ζωέ, ε, τα μέσα διαβίωση, που είναι ανοιχτή προ τον κόσμο αλλά μπορεί να φροντίσει τον εαυτό τη, που είναι ανθεκτική, πράσινη, ψηφιακή και που επενδύει στο μέλλον τη με όλες τις χώρες μαζί. Αυτό θα μας οδηγήσει στην ανάκαμψη. Θα είναι ένα μακρύ μονοπάτι, ένας δρόμος ε, τον οποίο θα πρέπει να βρούμε μόνοι μας. Η κρίση θα ανασχεδιάσει τις πολιτικές μας, τη γεωπολιτική μας κατάσταση, ίσως και την ίδια την παγκοσμιοποίηση. Και σε αυτόν τον νέο κόσμο η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη σε υπό οποιασδήποτε συνθήκε, όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες Και όταν κοιτάω στην ένωσή μα και βλέπω την ανθρωπιά, την ευρηματικότητα, ξέρω ότι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό και ότι ούτω και θα πράξουμε. Αξιότιμα μέλη λένε ότι μια ισχυρή ψυχή λάμπει πάντα μετά από οποιαδήποτε καταιγίδα. Εάν υποστηρίξουμε σήμερα την Ευρώπη με θάρρος, εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη, είμαι βέβαιη ότι αύριο η ψυχή της Ευρώπης θα λάμψει πιο φωτεινά από ποτέ. Ζήτω η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. για αυτό το στάδιο. Έχουμε και τη δυνατότητα να γίνουν και κάποιες συνδέσεις με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Ελπίζω να λειτουργήσει σωστά το σύστημα και να μας δοθεί η δυνατότητα να πειραματιστούμε και με νέους μηχανισμούς, οι οποίοι φυσικά είναι ακόμα ε, στο στάδιο του πειρασματισμού. Ο πρόεδρος Γκονζάλες Πόνς ε, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αγαπητέ Νταβίδ, αγαπητέ Σάρλ, αγαπητή Ούρσουλα, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να κλείνει το κοινοβούλιο, ε, δεν μπορεί να είναι κάτι απομακρυσμένο. Όπως ε, και τα σούπερ μάρκετ, όπως και οι πυροσβέστες, είμαστε και εμείς μια πολύ σημαντική λειτουργία. Είμαστε το νοσοκομείο της δημοκρατίας. Είμαστε εδώ σήμερα, αλλά εκατομμύρια συμπολίτε μας αναρωτιόνται πού ήμασταν όταν ξεκίνησαν όλα αυτά. Μετά το παράδειγμα τη. Ε, μετά από αυτό που είπε ο θέλω να το πω και εγώ. Μπορούσαμε να είχαμε δράσει νωρίτερα, να είχαμε δράσει καλύτερα και πιο ενωμένα. Και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό. Οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν φταίνε γι' αυτό που συνέβη, αλλά έπρεπε να, την, να το περίμεναν και έπρεπε να αντιδράσουν πιο γρήγορα. Και δεν κάναμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα ήταν καλό λοιπόν να ζητήσουμε συγγνώμη οι νεκροί ηλικιωμένοι άνθρωποι σήμερα είναι ήρωες πολέμου, είναι θύματα. Επιτρέπονταν από την κίνηση ένα δώσαμε σημασία. Και μπορεί να ξανακάνουμε αυτό το λάθος εάν θεωρήσουμε ότι αυτός ο εφιάλτης θα τελειώσει με το καλοκαίρι. Στην Ισπανία μάθαμε χθε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 νεκροί που δεν έχουν μετρηθεί. Οι περισσότεροι είναι οι ηλικιωμένοι που πέθαναν σε οίκους ευγυρίας. Και καθώς γίνονται όλο και περισσότερα τεστ, εμφανίζονται όλο και περισσότερα κρούσματα. Κάνουμε λάθο όταν θεωρούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα με τον ιό αυτόν. Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου το χειρότερο σενάριο. Ήδη κάνουμε σχέδια, λες και ο ιός δεν θα επανέλθει το φθινόπωρο. Και αν επανέλθει, λέμε ότι θα επανέλθει και θα είναι αποδυναμωμένος. Ή θα έχουμε ένα εμβόλιο. Και αν δεν το έχουμε, το, το 1918 το δεύτερο κύμα της γρήπης ήταν το χειρότερο. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη μπορεί να πλήρωσε, πλήρωσε το τίμημά τη, αλλά τι θα γίνει εάν υπάρξει έκρηξη στην Αφρική ή αλλού. Δεν λέω να σκεφτόμαστε μόνο το χειρότερο, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αποκλείουμε στου πολιτικοί θύνοντε. Στην Κίνα ξεκίνησαν όλα και είχαμε 3.300 νεκρούς. Στην Ισπανία, με 4% του πληθυσμού της Κίνας, έχουμε 18.000 και δεν του μετράμε καν όλους και στην Ιταλία 21.000 εάν λάβουμε υπόψη μα ότι η Ιταλία και η Ισπανία έχουν δύο από τα καλύτερα συστήματα υγεία στον κόσμο τι, σημαίνει, συμβαίνει τελικά η Κίνα μας έδειξε την αλήθεια τι παιχνίδι παίζουμε τελικά ο κορονοϊός η ανεργία ο εθνικισμός, λαϊκισμός και το ψέμα είναι τα τέσσερα κακά, οι τέσσερις πληγές αυτή τη στιγμή εδώ αυτή τη στιγμή αυτός ο ιός σκοτώνει τη γενιά των πατεράδων μας και έχουμε την εντύπωση ότι τα πράγματα συνεχίζονται όπως πάντα. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, πραγματικά η ενιαία αγορά είναι η πρώτη προτεραιότητά αυτή τη στιγμή. Κάποιοι έρχονται στι Βρυξέλλε για να δουν τελικά πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν. Κάποιοι άλλοι έρχονται στι Βρυξέλλε έρχονται επίση για να μην πάρουν άλλοι τα χρήματα. Κανεί όμω δεν ενδιαφέρεται για το σύνολο των Ευρωπαίων τελικά. Το να έρθει κάποιο στην Ευρώπη για να υπερασπιστεί μόνο τα, τα εθνικά του συμφέροντα και αυτό είναι εθνικισμό. Ακόμα και αν δεν το ξέρουν από ό,τι φαίνεται οι πρωθυπουργοί μα. Εάν ο, ο, ο φόβο για το θάνατο μα επηρεάζει όλου, αν ο θάνατο μα επηρεάζει όλου, εφόσον ο ιό δεν κάνει διαφορά από μια χώρα στην άλλη, γιατί οι εθνικέ κυβερνήσει να κάνουν αυτή τη διάκριση σε ό,τι αφορά του νεκρού ανάλογα με την εθνικότητά του. Δεν είμαστε τη στιγμή ε, που θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό η Κίνα έφτιαξε ένα νοσοκομείο πιο γρήγορα από ό,τι χρειάστηκε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συνέλθει το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο αποτελεσματική η διδακτορία τη Κίνα. Όχι, είναι ότι εμεί δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Πρέπει να δείξουμε ότι ο Ευρωπαϊσμό μπορεί να είναι και αποτελεσματικό, ότι ο Ευρωπαϊσμό μπορεί να είναι επικό, ότι μπορεί να είναι πατριωτικό, ότι ο Ευρωπαϊσμό μπορεί να είναι ανθρώπινο. Είναι η στιγμή να δείξουμε ότι τα σύνορα δεν θα είναι ποτέ λύση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια πανδημία που αφορά το σύνολο τη Υπήρου, τότε σε τι τι χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, ήρθε η ώρα, τώρα είναι η ώρα, ή τώρα ή ποτέ, στο ΕΛΚ, τα, στα άλλα κόμματα που, που, που υποστηρίξαμε, ψήφισαμε το ψήφισμα, κάναμε μια προσπάθεια συνένεση. Ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγάλη ελπίδα εκατομμυρίων Ισπανών που έχουν πληγεί ή που έχουν πεθάνει ή που είναι άρρωστοι από αυτό τον ιό δεν πρέπει να δώσουμε δίκιο στους λαϊκιστές, δεν πρέπει να δώσουμε δίκιο στους εθνικιστές, να μην δώσουμε δίκιο στους ψεύτες. Η ισπανική γρήπη σκότωσε κυρίως από πείνα και όχι από πυρετό. Μην δώσουμε λοιπόν τη νίκη στον ιό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα να δούμε αν θα μπορέσουμε να ακούσουμε την παρέμβαση της συναδέλφου Γκαρθία Πέρες. Θα συνδεθούμε μαζί της. Παρακαλώ, Ιράτσε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ ε, κύριε Σάσολη, κύριε Πρόεδρε, ε, κυρία Φοντερ Λάιεν, ε, κύριε Μισελ. Τα πρώτα λόγια που θα ήθελα να πω θα πάνε για τα θύματα αυτής της κρίσης και για όλους όσους οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή ή στα σπίτια τους προσπαθώντας να νικήσουν τον ιό και να ευχαριστήσω βεβαίως όλους τους επαγγελματίες που αυτές τις μέρες παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή του. Ξεκινώντα βεβαίω από το υγειονομικό προσωπικό, αλλά και τι δυνάμει ασφαλεία, ε, του ε, εργαζόμενου στα σούπερ μάρκετ, του μεταφορεί, του γεωργού, ε, αυτού που εργάζονται στου οίκου ευγυρία. Για όλου και όλε, διότι οι περισσότερε είναι γυναίκε από αυτού, εκατομμύρια, χιλιάδε ευχαριστώ. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ιστορία μα. Αυτή η πανδημία του κορονοϊού μα έχει χτυπήσει με έναν τρόπο που δεν μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί. Η ασφάλειά μας, η ελευθερία μας, η ελευθερία κίνησης, η καθημερινότητά μας δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα αλλάξουν και πώς θα είναι στο μέλλον. Ορισμένα πράγματα δεν τα ελέγχουμε. Κάποια άλλα όμως εξαρτώνται από εμά. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Οι αποφάσει που παίρνουμε σήμερα θα δείξουν κατά πόσο η Ευρώπη θα βγει ενισχυμένη ή κατά πόσο οι Ευρωπαίοι πολίτε θα χάσουν την εμπιστοσύνη του σε αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο. Είδαμε στην αρχή τη κρίση πω αυθόρμητα βγήκαν μπροστά οι εγωισμοί, οι εθνικισμοί. Σιγά σιγά καταφέραμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει και να βάλει μπροστά κάποια μέτρα αλληλεγγύης. Διότι γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε μετά το τέλος του, Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια στιγμή καταστροφής για να σταματήσει ο ανταγωνισμός μεταξύ των, των κρατών και έτσι ώστε η ανοικοδόμηση να φέρει ευημερία για όλους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίση που είναι συγκρίσιμη μόνο με τη μεγάλη κρίση ε, την προπολεμική. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο παρεμφερέ με αυτό του σχεδίου Marshall. Δεν αρκεί να αυξηθεί ο προπολογισμό. Πρέπει να υπάρχει μια πραγματική στρατηγική επενδύσεων και ενίσχυση των ε, στρατηγικών τομέων για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε το μέλλον τη Ευρώπη. Αυτή λοιπόν είναι η στιγμή που μπορούμε και πρέπει να φανούμε φιλόδοξοι, να ανοικοδομήσουμε την Ευρώπη πάνω σε μια νέα βάση. Αυτή η κρίση μας δείχνει τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν και τις ανισότητες μεταξύ των εδαφών, τις γεωγραφικές ανισότητες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή η κρίση να ανοίξει ένα ακόμα μεγαλύτερο χάσμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν δημόσιες πολιτικές για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα μπορούμε να προστατευτούμε το ίδιο. Δημόσιες πολιτικές λοιπόν, υγεία πρώτα απ' όλα, ε, να προστατεύσουμε τα εκατομμύρια Ευρωπαίους που χάνουν την εργασία τους, χάνουν τη δουλειά τους, δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα στο τέλος του μήνα, πώς θα πληρώσουν τον νίκη τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή οικονομία ισχυρή και αλληλέγγυα. Και θα πρέπει πλέον η Ευρωζώνη να έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει αυτές τις μεγάλες ε, χρηματοοικονομικές αλλαγές της παγκόσμιας. Θα πρέπει λοιπόν μέρος του χρέους ε, να ε, γίνει κοινό όπως προτείνουμε με αυτά τα ομόλογα της ανοικοδόμησης. Θα πρέπει επίσης η οικονομία αυτή να, είναι, να σέβεται περισσότερο το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους να είναι πιο ψηφιοποιημένοι. Αυτή η κρίση μα δείχνει ότι είναι αναγκαίο να εκδημοκρατήσουμε την τεχνολογία, έτσι ώστε όλοι οι πολίτε, όλε οι επιχειρήσει, όπου και αν βρίσκονται, να μπορούν να υποφελθούν από αυτήν για την εργασία, για τι σπουδέ, για την έρευνα, για τι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων. Βλέπουμε αυτέ τι μέρε πω πολλά παιδιά που επειδή δεν έχουν πόρου, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα επιγραμμικά θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Όλες αυτές οι ιδέες δεν είναι καινούριε. Ε, υπάρχουν στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό. Το πράσινο deal, τα ευρωομόλογα, το συζητούσαμε ήδη το 2008 αυτό. Όμως είναι πιο επίγον από ποτέ να προχωρήσουμε. Είναι η ώρα της αλήθειας. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ε, να μην είμαστε εκεί στο ραντεβού με την ιστορία. Το είπαμε και στο κοινό μας ψήφισμα, το οποίο μπορούσαμε να αντιπραγματευτούμε μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα βεβαίω ε, να είχαν συμμετάσχει και άλλε ομάδε. Ελπίζω οι βουλευτές και άλλων ομάδων, πολιτικών ομάδων να έρθουν ε, να συμμετάσχουν σε αυτή την έκκληση την κοινή του Κοινοβουλίου έτσι να δράσει η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ξέρουμε τι πρέπει να συμβεί. Χρειάζεται απλά το πολιτικό θάρρο για να προχωρήσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύει ότι σήμερα έχουμε καταλάβει τις ιστορικές μας ευθύνες. Έχουμε αντιληφθεί ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις ιδεολογικές ε, εθνικές ε, διαφορές μας για να σκεφτούμε το κοινό συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Σε αυτό το ψήφισμα προτείνουμε επίγοντα μέτρα και κάποια άλλα πιο μεσομακροπρόθεσμα. Όλα αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα. Τα επίγοντα για να σώσουμε ζωές αλλά και για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ένα δίχτυ προστασία που χρειάζονται τόσοι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όσο περισσότερο δράσουμε και πιο γρήγορα δράσουμε σήμερα, τόσο μικρότερο θα είναι ο αντίκτυπο ε, τη οικονομική κρίση στο μέλλον, τόσο πιο γρήγορα θα, έρθει η ανάκαμψη και θα επανέλθει μια κάποια κανονικότητα. Σε μια στιγμή ενότητα και συνεργασία, τη διεθνού συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε την απόφαση του Τραμπ ε, να διακόψει τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. και θα πρέπει και εμεί στην Ευρώπη το θέμα αυτό να το δούμε. Πρόκειται και μια κρίση που αφορά όλε τι χώρε τη Ένωση, που τι πλήττει όλε. και θα πρέπει όλε οι χώρε να βγουν από την κρίση αυτή εξίσου ισχυρέ και εξίσου αποφασισμένε. Θα ήταν απαράδεκτο ο COVID-19 να δημιουργήσει νέε ανισότητε μεταξύ κρατών μελών καθιστρώντας ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή σύγκληση πολλοί πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν απογοητευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως σημαίνει ότι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν απογοητευτεί επειδή ελπίζουν περισσότερα από εμά. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να αποδείξουμε ότι αξίζει τον κόπο να πιστεύει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι οι αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης που αναφέρουμε και, και λέμε είναι αληθινέ, αληθινές και ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε αυτό. Εάν το Συμβούλιο, εάν η Κομισιόν δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων στην αρχή της κρίσης, το Κοινοβούλιο θα απαιτήσει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τώρα, δεν είναι αργά. Έχουμε ένα μακρύ δρόμο μπροστά μας. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου πρέπει να γνωρίζουν ότι χρόνος υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Είναι δική μας ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ την Πρόεδρο Γκαρσία Πέρες και τώρα ο Πρόεδρος Τσόλος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.